διότι οι γραπτές δηλώσεις είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε. Πρόεδρος, πάμε τώρα στη ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την έκθεση Μπέρες. συγγνώμη, λέει ο της κυρίας Μπερές για την τροποποίηση του κανονισμού 1927 που δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην ε, Παγκοσμιοποίηση. Ε, λοιπόν, υπέρ, γιατί κατά αποχές εγκρίνεται και το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξης ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται σαφώς. Επόμενο θέμα είναι έξι προτάσεις ψηφίσματος για την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Έχουμε κοινή πρόταση ψηφίσματος και ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και συγχαρητήρια. Επόμενο θέμα, πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά την Σύνοδο Κορυφής γύριο ε, του Ρίου, συν 20. Ξεκινάμε την παράγραφο 4, υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος, ε, έναρξη ψηφοφορίας, λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 19, σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, τι περιπτώσει καταπίπτει. Παράγραφος 6, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 8, έχουμε προφορική τροπολογία του κυρίου Λάινεν, Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά την παράγραφο 8, διότι η διατύπωση είναι παραπλανητική. Λέει στο παλιό κείμενο ότι ανησυχεί, διότι εστιαζόμεθα στην πράσινη οικονομία και θεωρείται ένα από τα δύο βασικά θέματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο, δίνει αρνητική χρειά το ότι ανησυχεί, που αφορά το, το ότι τονίζεται η πράσινη οικονομία σαν ένα από τα δύο θέματα. Όχι is concern, αλλά concerning. Όχι ότι ανησυχούμε, αλλά ότι αφορά. Αυτό. Αυτή είναι η εξήγηση προς τους πρασίνους που με ρώτησαν είναι θετικό, θετική διατύπωση, αρνητική. Είναι θετική. Πρόεδρος, όλοι καταλαβαίνουν. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 24, τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος, αν θέλετε έλεγχο, ας κάνουμε τον έλεγχο. Έλεγχο στην τροπολογία 16, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λήξεις. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται σαφώς, συνάδελφοι. Παράγραφος 25, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τρίτο τμήμα, υπέρ, τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, αυτή τη φορά πρέπει να γίνει ο έλεγχος, Έλεγχο για το τρίτο τμήμα της 25 έναρξης ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα... We have amendment number 12. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Καλός έλεγχος για την τροπολογία 4 έναρξης. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της παραγράφου, υποφάτα παράγραφου 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφο 29 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία έναρξη ψηφοφορίας λήξεις εγκρίνεται Τρίτο τμήμα. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξης ελέγχου για το τρίτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Παράγραφος 34, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται cloud. Τέλος πληροφορίας Και εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 τώρα. Όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 38. Σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 13. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στο αρχικό κείμενο στο εδάφιο 39. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Όχι ακόμα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα είχατε χρόνο να ψηφίσετε όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα επισημαίνεται κάτι στον Πρόεδρο εκτός μικροφώνου. Φοβούμαι ότι θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όπως μπορείτε να δείτε στις οθόνες ακόμα έδειχνε άλλη τροπολογία. Τροπολογία 13. Ψηφίζουμε όμως το εδάφιο 39, το αρχικό του κειμένου 39. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά για το 39. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 39, εδάφιο 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπομονή, συνάδελφοι, παρακαλώ. Άρχεται λοιπόν τώρα η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και εγκρίθηκε. Τροπολογία 6, εδάφιο 40. Όσοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε στην 40 σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Τη 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα. Εδάφιο 40. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Και τροπολογία 14. <clears throat> Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 24 τώρα. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και έτσι περνάμε τώρα στο εδάφιο 47 σε τμήματα ψηφοφορία, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Δεν ξέρω τι γίνεται στην αριστερή πτέρυγα, όπως βλέπω εγώ αν ψηφίζεται υπέρ ή κατά. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Όσοι είσαστε υπέρ, σηκώστε τα χέρια. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα. Εδάφιο 47. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και πάλι η ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το τρίτο τμήμα του 47. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα στη συνέχεια η τροπολογία 9 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Πάμε κατευθείαν στην τροπολογία 23. Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος εδάφιο 50 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα του 50 ψηφίζουμε. Άρχεται. Δεύτερο του 50. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Εδάφιο 54. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Παράγραφος 59. Όσοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Λυπούμε που πρέπει να σας ενοχλήσω, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Εδάφιο 60 σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστικά, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε και αυτό. Εδάφιο 61. Όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το 61. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Εδάφιο 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή τη φορά νομίζω ότι απορρίφθηκε και μπορώ να το πω αυτό. Τελεσίδικα. Να ελέγξουμε. Εντάξει, πολύ ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Αφού το ζητήσατε θα ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίθηκε βλέπετε. Τροπολογία 21 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Εδάφιο 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το 67. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 17. Υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Και τώρα εδάφιο 71. Έχουμε σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 15 <clears throat> με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Εδάφιο 80. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αλλά θα έλεγα για να γνωρίζουμε το ακριβές αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Παράγραφος εδάφιο 87. Τροπολογία 22 επ' αυτού. Όσοι είσαστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Εδάφιο 89. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Εδάφιο 93. Και πάλι ονομαστικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αυτή τη φορά αυτό απορρίφθηκε. Εδάφιο 96 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι ακόμα, εντάξει, όχι ακόμα. Συνεχίζεται η ψηφοφορία, άρχεται και συνεχίζεται η ψηφοφορία. Τώρα λίγη η ψηφοφορία. Και το αποτέλεσμα είναι απορρίφθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. <clears throat> στο K έχουμε δύο τμήματα. Με ονομαστική ψηφοφορία το πρώτο, άρχεται η ψηφοφορία από αυτού. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα σαφώς εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα και πάλι ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε και αυτό με μικρή διαφορά αλλά εγκρίθηκε εν πάση περιπτώσει. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και με σαφές αποτέλεσμα εγκρίθηκε σαφώς συγχαρητήρια. Now we will vote on the... Τώρα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα της Επιτροπής Απασχόλησης όσον αφορά το μέλλον του Ταμείου για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Τροπολογία αριθμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την παράγραφο 5 την αρχική υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της, τροπολογ... της παραγράφου 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 δέλτα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι πεπισμένος στη ψηφιζική το κέντρο. Ξανά λοιπόν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το επόμενο ψήφισμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τέλος, έχουμε την τελευταία για σήμερα ψηφοφορία που είναι το ψήφισμα του κύριου Νταφ και άλλων σύμφωνα με το άρθρο 96 της ε, ε, διαδικασία όσον αφορά το πρωτόκολλο συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της Ελία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου. Το λόγο έχει ο κύριος Νταφ. Παρακαλώ, κύριε Νταφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα θέλει το πρωτόκολλο αυτό να εξεταστεί και πάλι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά τη συμβατότητά του. Θέλουμε γνώμη δηλαδή του δικαστηρίου. Πρόκειται για μια δοκιμή όσον αφορά τη συμβατότητα της συμφωνίας με την συνθήκη όσον αφορά το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. τα αποτελέσματα δεν είναι να αρθεί η τρέχουσα συμφωνία. Η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο. Το Κοινοβούλιο πάντως οφείλει να φροντίσει για τη συμμόρφωση στη συνθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάφ. Ψηφίζουμε λοιπόν το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα που είχαμε να ψηφίσουμε για σήμερα. Έχω βέβαια κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω στα τσεχικά, λέει ο Πρόεδρος. Έχω λάβει τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την πρώτη ανάγνωση ε, τις ε, αιτιολογήσεις ε,